η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12. Και τώρα... Τώρα και κύριοι να περάσουμε στο επόμενο σημείο, προφορική ερώτηση στην Κομισιόν Αντίκτυπο των Μέτρων Λιτότητα Συνθήκε Ζωή των Ανθρώπων με Αναπηρία. Πρώτα θα πάρει το λόγο η κυρία Περβάνς Περές. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συναδελφοί. Η Επιτροπή Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων ε, ήθελε να θέσει την Ολομέλεια το θέμα του αντικτύπου των μέτρων λιτότητα στι συνθήκε ζωή ε, των ανθρώπων με αναπηρία. Και πριν να σα παρουσιάσω αυτή την προφορική ερώτηση, να σας πω ότι προδήλως ε, Εκτός ε, του δικού μας ε, οίκου υπάρχει πολύ μεγάλη απήχηση. Ε, υπήρξαν πάρα πολύ σημαντικές αντιδράσεις σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις και σε διάφορους φορείς που ασχολούνται με τους ανθρώπους με αναπηρία και ανησυχούν για τη μοίρα τους. Όταν ένας άνθρωπος στους 10 είναι ανάπηρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και το ποσοστό της φτώχειας των ανθρώπων αυτών είναι άνω του 70% σε σχέση με το μέσο όρο του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, υπάρχει μόνο 45% των ανθρώπων αυτών που απασχολούνται μόνο το 25% γνωρίζει ένα πρόβλημα ε, ψυχικής υγείας ε, και πολλοί από αυτούς μπορεί να οδηγηθούν ε, σε αναπηρία. Πάνω από 20% των ανθρώπων αυτών πάσχουν από βαριές αναπηρίας Έχουμε 35% προβλήματα μάθησης ε, σε ανθρώπους ε, με βαριά αναπηρία ε, έτσι λοιπόν αυτό είναι το διακύβευμα του θέματος που θέτουμε εδώ. Ξέρουμε όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα οπλοστάσιο για το οποίο είστε υπεύθυνοι κυρία Επίτροπε ε, σε σχέση και με τη χάρτα των Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων καθώς ε, λέγεται ότι είναι απαραβίατη ανθρώπινη αξιοπρέπεια στο άρθρο 1 και στο άρθρο 21 λέγεται ότι οι διακρίσει κατά την ανθρώπων ομοιρία αντίκειται στο δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στο άρθρο 26 αναγνωρίζεται το δικαίωμα ε, των ανθρώπων με αναπηρία ε, να επωφελούνται από μέτρα που διευκολύνουν, πρέπει να ωφελούνται οι άνθρωποι αυτοί από μέτρα που διευκολύνουν τη συμμετοχή του στην κοινωνική ζωή. Δεν θα αναφερθώ ούτε στην συνθήκη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στη Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών, αλλά θα ήθελα να απευθυνθώ στην Κομισιόν ε, για τι προτεραιότητας στρατηγικής 2010-2020 ε, είχε δηλώσει την πρόθεση να εγγυηθεί στου ανθρώπου με ανεπηρία την πρόσβαση στα αγαθά και στι υπηρεσίε και στις δημόσιε υπηρεσίε και σε μηχανισμού βοήθεια. Ενώ στην ίδια η Κομισιόν ανέφερε ότι θα έπρεπε να πράξουμε έτσι ώστε οι άνθρωποι με ανεπηρία να συμμετέχουν πλήρω στην κοινωνική ζωή, ε, παρέχοντας υπηρεσίες εγκύτητας, ποιοτικέ ε, και ε, πρόσβαση σε προσωπική βοήθεια. επίση ανέφερε ότι θα πρέπει να επιτραπεί στου ανθρώπου με ανεπηρία να έχουν αξιοπρεπέ εισόδημα, να εργάζονται στην κανονική αγορά εργασία. Αντέδρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μια έκθεση του κυρίου Κόσα σε ένα ψήφισμα 25 Οκτωβρίου 2011. Σήμερα τι διαπιστώνουμε όμως. Διαπιστώνουμε ότι οι πολιτικές λιτότητες επιδεινώνουν ε, την ήδη πολύ δύσκολη κατάσταση των ανθρώπων ε, με αναπηρία Μειώνοντα ε, τι δημόσιε δαπάνε, στον τομέα τη υγείας και τη ε, πρόσβαση στη φροντίδα, στην περίθαλψη, περιορίζοντα τι επενδύσει στι ε, βασικέ δομέ, την κινητικότητα και για τη συμπερίληψη των ανθρώπων με αναπηρία. Οι στόχοι τη στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση 2020 συνιστούν στο να φτάσουμε σε ένα ποσοστό απασχόληση 70% από τους άτομα 25 60 και να μειωθεί η ανεργία στους ανθρώπους που απειλούνται ε, με αποκλεισμό. Αν δεν ε, εντάξουμε τους ανθρώπους με αναπηρία στην αγορά εργασίας, τότε δεν θα πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Πέραν αυτού το διακύβημα είναι την ίσον ε, ευκαιριών για μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία διέπεται από τις αρχές της ισότητας και πρέπει να προσφέρει στους ανθρώπους με αναπηρία τις ευκαιρίες να ελοποιήσουν τα σχέδια στη ζωή τους ε, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξέρει να δράσει για τους ανθρώπους με αναπηρία. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απαραίτητο να ε, είναι συνεκτική με την στρατηγική που ίδια υιοθέτησε και που υποστήριξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε αυτή τη δράση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει ίσως να αποσαφηνίσει τι δράσεις θα μπορούσε να βάλει σε εφαρμογή Κομισιόν. Επίσης ζητάμε από την Κομισιόν να δηλώσει διαθεσιμότητα για να εξετάσει αυτό που θα εκπονήσει ως πρόταση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως πρόταση σύστασης βάσει της έκθεσης που εκπονεί τώρα η κυρία Λάμπερτ ε, για την ε, ε, πρόσβαση των ευάλωτων πληθυσμών στο σύστημα υγείας. από μένα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και θα ζητήσω από την Επίτροπο Ρέντινγκ να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω προς την εισηγήτρια ότι το μήνυμά της το ακούσαμε και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει πολύ προσεκτικά όχι μόνο αυτά τα οποία προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και αυτά τα οποία θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι το ίδιο επιθυμούμε. Θέλουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών ή αδίποτε θεμελιώδη δικαιώματα να γίνονται σεβαστά. Και διαβεβαιώνω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι φέτος θα προχωρήσουμε με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την προσβασιμότητα, για το accessibility, πράγμα το οποίο έχουμε υποσχεθεί. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία και ε, θα προχωρήσει. Συμφωνώ με την εισηγήτρια όταν λέει ότι η γύρανση του πληθυσμού και η οικονομική κρίση, γιατί και τα δύο συνδυάζονται, ότι πιέζουν το σύστημα κοινωνικής προστασίας. Η χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών γίνεται όλο και πιο δύσκολη και ταυτόχρονα γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι απαραίτητο να βρεθούν ε, νέα ενάψματα για την ανάπτυξη και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία η απασχόληση όλων των τομέων του πληθυσμού και εδώ συμπεριλαμβάνω και τα ποσοστά απασχόλησης των ατόμων με αναπηρίες. Επίσης γνωρίζουμε όλοι ότι τα άτομα με αναπηρίες αντιμετωπίζουν περισσότερους φραγμούς από ότι τα υπόλοιπα τμήματα του πληθυσμού. Αυτό ισχύει και σε εποχές ανάπτυξης της οικονομίας. Φανταστείτε λοιπόν πόσο πιο δύσκολο είναι σε περίοδο κρίσης. Οι λιγότερο εκπαιδευμένοι και οι φτωχότεροι Ευρωπαίοι βρίσκονται σε ακόμη χειρότερη κατάσταση σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Ορισμένες ομάδες πολιτών γίνονται όλο και περισσότερο ευάλωτες και διατρέχουν τον κίνδυνο αποκλεισμού σε μεγαλύτερο βαθμό. Μια πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού ε, Ιδρύματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αναπηρία ε, τονίζει ότι η μείωση των δαπανών για τις κοινωνικές υπηρεσίες ε, μπορεί να καταλήξει σε δυσανάλογη αύξηση των ατόμων με αναπηρία που χάνουν τη θέση εργασίας τους. Δεν είναι λοιπόν μια οριζόντια σχέση, αλλά μια γεωμετρικά αυξανόμενη σχέση και πραγματικά φύγεται αυτό το τμήμα του πληθυσμού σε μεγαλύτερο βαθμό. Εξετάσαμε έξι κράτη-μέλη, Ιρλανδία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία και Ηνωμένο Βασίλειο. Κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου υπάρχει οικονομική κρίση και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αγνοήσει αυτή την εκθετική ανάπτυξη των ατόμων με αναπηρία. Κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, οι συστάσεις για την Εσθονία, τη Δανία και την Ολλανδία ε, παραθέτουν θέματα που έχουν σχέση με την αναπηρία στα υπηρεσιακά έγγραφα. Όπως θα γνωρίζετε, η Επιτροπή ασχολείται τώρα με τις συστάσεις για τον ε, κύκλο του 2013 και νομίζω ότι δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση, το αντίθετο μάλιστα. Πιστεύουμε ότι η αναπηρία είναι ένα θέμα που περνάει σε όλους τους τομείς και καταβάλουμε μια πραγματική προσπάθεια να συμπεριλάβουμε το πρόβλημα αυτό, να συμπεριλάβουμε την πραγματικότητα αυτή σε όλες τις πολιτικές μας. Στην Ευρώπη του 2020 και στη στρατηγική ανάπτυξη θέλουμε να συμπεριλάβουμε ε, πολιτικές για την αναπηρία. Και το πακέτο για τις κοινωνικές ε, επενδύσεις ε, απαιτεί να, συμμετέχουν τα κρατημέλη σε επενδύσεις που θα βελτιώνουν τις ικανότητες των πολιτών να αντιμετωπίζουν ε, τον κίνδυνο. Και γι' αυτό οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου μιλούν για πρόσβαση σε προσιτές υπηρεσίες ποιότητας συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγείας ε, γενικού ενδιαφέροντος και αυτό είναι μία από τις έξι προτεραιότητες για τις επενδύσεις και συμπεριλαμβάνεται και η ανάπτυξη ε, ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας που θέλουν να αποφύγουν ε, την ε, ιδρυματοποίηση, γιατί και η ιδρυματοποίηση είναι άλλο ένα πρόβλημα το οποίο πολλές φορές έχουμε συζητήσει στο παρελθόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και υπάρχει μία λογική της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Και ζητώ συγγνώμη που μιλώ για τη λογική της οικονομίας, αλλά και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη, διότι εδώ υπάρχει μία πιθανότητα ανάπτυξης ορισμένων τομέων της ε, κοινωνικής οικονομίας. Θα ήθελα να αναφέρω, παραδείγματο χάρη, τι θέσει εργασία στον τομέα τη υγεία και τη περίθαλψη. Είναι ένα τομέα όπου μπορούμε να έχουμε αύξηση των θέσεων εργασία. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω και τις θέσεις εργασίας στην πράσινη οικονομία, τις θέσεις εργασίας στην ψηφιακή οικονομία. Εδώ υπάρχει πραγματικά δυνατότητα ανάπτυξης και αυτό είναι κάτι που έχουμε εντοπίσει στις, στην ετήσια μελέτη για την ανάπτυξη το 2012, όπου η Επιτροπή συνιστά τα κράτη-μέλη να λάβουν πρωτοβουλίες για να διευκολύνουν την ανάπτυξη αυτών των τομέων και των αντίστοιχων των θέσεων εργασία. Θα σα δώσω αριθμητικά στοιχεία για τι αποκαλούμενε λευκέ θέσει εργασία, στην υγεία και περίθαλψη. 22 εκατομμύρια άτομα εργάζονται το 2010 σε αυτό το τομέα, 1,5 εκατομμύρια περισσότερα αναμένονται μέχρι το 2020 και θα αποτελούν το 10% της συνολικής απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών αντιστοιχούν στο 5-13% του ΑΕΠ και προσφέρουν 800 εκατομμύρια ετησίως ως κύκλο εργασιών στην ευρωπαϊκή οικονομία. 800 δισεκατομμύρια, συγγνώμη. Υπάρχει μεγάλη πίεση όσον αφορά τους μισθούς ε, σε αυτόν τον τομέα της υγείας ε, και των κοινωνικών υπηρεσιών, αυτών των λευκών θέσεων εργασίας. Παρ' όλα αυτά πρέπει να εξετάσουμε αυτούς τους τομείς για να δούμε πώς μπορούμε ε, να αναπτύξουμε τον τομέα και τις θέσεις εργασίας και τις θέσεις εργασίας γύρω από την ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Θα πρέπει να εξετάσουμε και τις φορολογικές πολιτικές διότι σε πολλά κράτη-μέλη μπορεί να υπάρχουν και υπάρχουν φορολογικά κίνητρα για να ε, δοθεί δυνατότητα στις εταιρείες να προσλάβουν άτομα με αναπηρία και για να μπορέσουν τα άτομα με αναπηρία να μπουν ή να επανέλθουν στην αγορά εργασίας. Και αυτό με φέρνει στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία γιατί οι περισσότερες δράσει για τον τομέα αυτό ξεκινούν από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και εδώ έχουμε μια οδηγία του Συμβουλίου του 2007-2008 ένα γενικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση. Έχει μεταφερθεί σε εθνικό δίκαιο σε όλα τα κράτη-μέλη και είναι υπεύθυνα τα κράτη-μέλη για την υλοποίηση αυτού του νομοθετικού κειμένου. Η Επιτροπή απλώς μπορεί να παρακολουθεί το πώς εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη αυτή την οδηγία του Συμβουλίου στο εθνικό τους δίκαιο. Το 2013 θα συντάξουμε και μία έκθεση για την υλοποίηση αυτής της οδηγίας και την έκθεση αυτή θα τη συζητήσουμε βέβαια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να αναφερθώ και στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών ε, για τα άτομα με αναπηρίες. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέλος αυτής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών και εγώ πάντοτε πιέζω τα κράτη-μέλη ε, να προσυπογράψουν αυτές τις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Και φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει την πρώτη της έκθεση προς την Αρμόδια Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για το πώς εκπληρεί τις υποχρεώσεις της η Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με αυτή τη σύμβαση. Και ταυτόχρονα θα, αναθεωρήσουμε, θα επανεξετάσουμε την πρόοδο που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία που ανέφερε και η συγγήτρια και κατά τα μέσα του έτους θα έχουμε και ένα νομικό πλαίσιο για την προσβασιμότητα κάτι εξαιρετικά σημαντικό όχι μόνο για του, τα άτομα με αναπηρία αλλά ε, και για τους, ε, τα αυξανόμενα άτομα μεγάλης ηλικίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πίτροπε για τη λεπτομερέστατη αυτή ανάλυση. Να σας πω ότι εδώ μπροστά μου βλέπω ότι είχατε το λόγο κανονικά για τρία λεπτά. Γι' αυτό καμιά φορά έχουμε κάποια προβλήματα και πιέζω τους συναδέλφους για να μιλάνε λιγότερο. Απλώς μια παρατήρηση είναι αυτή, έτσι, ευχαριστώ. Για δύο λεπτά, ο κύριος Κόσα έχει το λόγο. Η κυρία Κόσα. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Ρέντινγκ, θα προσπαθήσω να είμαι απόλυτα συγκεκριμένος. Ε, χαίρομαι που γίνεται αναθεώρηση της ε, πολιτικής ε, για την αναπηρία και θα πρέπει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετάσχει. Γνωρίζουμε ότι η κατάσταση των ατόμων με αναπηρία σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδεινώνεται. Σήμερα φτάνει σε κατάλληλη χρονική στιγμή η συζήτηση. Θέλουμε να έχουμε θετικά πρότυπα, θέλουμε να έχουμε μακροπρόθεσμες στρατηγικές. Ε, να συζητήσουμε παραδείγματος χάρη τη στρατηγική της ε, Ουγγαρίας. Να συζητήσουμε το θέμα των Ινστιτούτων ε, για τα άτομα με αναπηρία. Πρέπει να καταβάλουμε ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες, ιδίως για τα άτομα αυτά τα οποία έχουν σοβαρές αναπηρίες. Θα πρέπει να δίδονται ευκαιρίες απασχόλησης και για τα άτομα με σοβαρές αναπηρίες. έχουν ε, καταργηθεί πολλές θέσεις ε, προστατευόμενης εργασίας για άτομα με αναπηρία και από την κατάργηση αυτών των θέσεων έχουν μείνει εκτός αγοράς εργασίας πολλά άτομα με αναπηρία. Πρέπει ε, να έχουμε υπηρεσίες που να προσφέρονται βάσει των αναγκών των ατόμων με αναπηρία και θα πρέπει να φροντίζουμε την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία που θα πρέπει να ξεκινά ήδη από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Να υποστηρίζουμε την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε θέσεις εργασίας γιατί για όποιον για ό,τι και να συζητάμε, ε, η προσβασιμότητα είναι πάρα πολύ σημαντική για οποιαδήποτε θέση εργασίας. Ακόμη θα ήθελα να πω ότι στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, δόθηκαν 700 δισεκατομμύρια για την ε, εξισορρόπηση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ε, και ε, τώρα βλέπουμε ότι έχουν μείνει στο δρόμο 270.000 άτομα με ε, νοητική καθυστέρηση. Το πιο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να εντάξουμε τα άτομα με αναπηρία στις πολιτικές μας και στην κοινωνία μας. Ευχαριστώ πολύ. Για δύο λεπτά η κυρία Γκάνς έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ συζητήσαμε πολύ τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και είπαμε ότι κυρίως τα άτομα με μεγαλύτερη ανάγκη πλήττονται από την οικονομική κρίση. Η προστασία των ατόμων με αναπηρία είναι σημαντική και θα πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το 2020. Η περικοπή των δημοσίων δαπανών δεν θα πρέπει ε, να αφήνει έξω από την αγορά εργασίας τα άτομα με αναπηρία. Στην ε, Ουγγαρία ε, μειώθηκε αναδρομικά η αναπηρική σύνταξη και τα άτομα αυτά των οποίων μειώθηκε η αναπηρική σύνταξη είναι άτομα που έμειναν χωρίς κοινωνικές παροχές. Θα πρέπει να επανεξεταστεί λοιπόν η διακριτική μεταχείριση ε, έναντι των ατόμων με αναπηρία ε, ε, που προκύπτει από την περικοπή των δαπανών και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προς αντιστάθμιση αυτών των προβλημάτων. Ευχαριστώ. Ξανά για δύο λεπτά η κυρία Άρκιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε, πρόσπατη διάσκεψη για άτομα με αναπηρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συνάδελφό μου, η Βάλερη Μόν, που είναι μάνατζερ του Κέντρου Ανεξάρτητη Διαβίωση στο Λόγκφορ στην Ιρλανδία, το είπε απλούστατα. Είπε άτομα με αναπηρία είναι πάντα σε περισσότερο κίνδυνο από τη φτώχεια και είναι πιθανότερο να ζουν σε φτώχεια. Όμω, σε ένα καθεστώ λιτότητα δεν έχουν καμία τύχη. Και γι' αυτό έχουμε αυτό το ερώτημα που βάλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι το αντίκτυπο στου απλού πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ενώση που ζουν σε καθεστώ ε, λιτότητα είναι πολύ ε, μεγάλο αντίκτυπο, αλλά είναι πιο σοβαρά τα πράγματα σε άτομα με αναπηρία. Και αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κάτι μελη θα πρέπει να κινηθούν ενεργά του να εξασφαλίσουν ότι εκείνοι που έχουν μια αναπηρία ε, δεν θα περιθωριοποιηθούν παραπάνω. Και πραγματικά για αυτού του λόγου η Επιτροπή Απασχόληση ζήτησε να υπάρξουν κοινωνικοί δείκτε δίπλα στου οικονομικού δείκτε στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Κατά τα τελευταία χρόνια στην Ιρλανδία είδαμε περικοπές στους αφορά υπηρεσίε και ώρες προσωπικών βοηθών και επιδόματα κινητοποίησης. Αυτό επέτρεπε σε άτομα που δεν μπορούσαν να περπατήσουν έχουν κάποια δυνατότητα να διαδράσουν κοινωνικά και ακόμα και να πάνε στη δουλειά. Και τώρα πολλοί κόσμος κινδυνεύει να είναι φυλακισμένο στο σπίτι του. Ο ε, πραγματικός μου φόβος όλα αυτά είναι ότι θα καταστρέψουμε πολλά χρόνια καλής δουλειάς και θα καταστρέψουμε ή θα αποδυναμώσουμε σημαντικά πολιτικές ένταξεις και δομές που οικοδομήσαμε με κόπους. Ο μεγαλύτερος μου πόλος επικεντρώνεται επί διαφόρων θεμάτων. Πρώτα απ' όλα, άτομα με αναπηρία θα ειδωθούν σαν ένα βάρος όσον αφορά το κράτος και σε πρόσφατη συνεδρίαση στην Επιτροπή απασχόλησε ένας εκπρόσωπος από το Βέλγιο ανα, αναφέρθηκε για την οτροπία που επικρατεί και περισσότερο. Δηλαδή ένα άτομο σε μια αναπηρική ελληνική πολυθρόνα είναι μια ευθύνη, ένα βάρο. Παίρνει τα χρήματά μου. Τα χρήματα του φορολογουμένου. Αυτό είναι συχνά ένα σχόλιο που ακούγεται. Δεύτερον, μετακινούμεθα από το μοντέλο κοινωνική ένταξη ιατρικό μοντέλο. Τρίτον, ε, οι θεράποντε, εκείνοι που παρέχουν ε, βοήθεια και οι οικογένειε ε, έχουν, έχουν προβλήματα. Η μείωση των υπηρεσιών και η ανεργία των ατόμων αναπηρία θα οδηγήσει σε όλο και περισσότερου ανθρώπου με αναπηρία που τελικά δεν μπορούν να βρουν δουλειά και ζουν στη φτώχεια. Για ένα λεπτό το λόγο έχει η κυρία Λαμπέρ τώρα. Ευχαριστώ. Καλωσορίζω την δυνατότητα να θέσουμε αυτά τα ερωτήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γνωρίζουμε πολύ καλά στο Κοινοβούλιο για την ανεργία που υφίσταται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά βεβαίω οι νέοι με αναπηρίε πιθανότατα θα έχουν τη μεγαλύτερη δυσκολία από όλου για να βρουν μάλιστα την πρώτη τους δουλειά ε, σε οποιοδήποτε τομέα, ακόμα και σε νέου τομεί. Λοιπόν, η πρόταση προσβασιμότητα που ανέφερε η Επίτροπο ήταν κάτι ευπρόσδεκτο. Επίση, θα θέλαμε να δούμε πραγματικά στεναρά ενεργό εφαρμογή των οδηγιών κατά πολέμηση των διακρίσεων που ήδη βρίσκονται ε, κατατεθειμένες και εφαρμόζονται. Οι περικοπέ, όπω γνωρίζουμε μειώνουν τι δυνατότητε για ανεξαρτησία και κοινωνική ένταξη ακόμα και σε χώρες που ήταν οι προδευτικότερες. Και πράγματι, όπω η Μάριον Χάρκιν, η συνάδελφο, είπε, όλο και περισσότερε ενδείξει δείχνουν ότι οι άνθρωποι με αναπηρία αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη εχθρότητα σε κάποια κράτη-μέλη. Πρόσφατη δημοσκόπηση τη οργάνωση οργάνωσης του Ηνωμένου Βασιλείου έδειξε ότι δύο τρίτα από εκείνους ε, που ρωτήθηκαν είχαν εμπειρία εχθρότητα ε, πάνω από 40% που ήταν εδώ και τέσσερι μήνε. Και αυτό αναφέρθηκε και στον τύπο, ακόμα σε ποιοτικό τύπο όπω είναι η Daily Telegraph. Είδαμε πρόσφατα ότι η βραχυπρόθεσμη οικονομική αντιμετώπιση θα έχει φρικτές μακροπρόθεσμες συνέπειες. Ευχαριστώ για 1,5 λεπτό. Ο κύριο Μέρφυ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πήρα την πρωτοβουλία μαζί με πολλέ ομάδε ή άτομα αναπηρία να προωθήσω αυτή τη συζήτηση ώστε να τονίσουμε την ομή, τη βίαιη πραγματικότητα που επιβάλλουν οι πολιτικέ λιτότητε που επηρεάζουν δυσανάλογα αυτού που έχουν αναπηρία, υψηλότερα επίπεδα ανεργία, περικοπέ, ζωτικών υπηρεσιών και περικοπέ όσον αφορά την εξάρτητη διαβίωση. Πολλά πολλέ περικοπέ έγιναν στην Ιρλανδία, τεράστιε περικοπέ όσον αφορά την προσωπική βοήθεια και αρρωγή και μείωση του επιδόματος κινητικότητας. Αυτές οι πολιτικές λιτότητες είναι πάνω από κάτι από δυσκολία, παραβιώζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά την απόψή μου. Τα δικαιώματα, το κίνημα για τα δικαιώματα κινητικοποίησεως κινήθηκε για σεβασμό όσον αφορά τη μετώπιση αυτών των τόπων και την αξιοπρέπεια. Είχε πολεμήσει να υποστηριχθούν τα άτομα με αναπηρία, ώστε να συμμετέχουν πλήρω στην κοινωνία και θα πρέπει να έχουν τα βασικά του δικαιώματα. Δικαίωμα να δουλεύουν, να μεγαλώσουν οικογένειες, δικαίωμα να εκπαιδευτούν αυτοί οι άνθρωποι. Όλα αυτά απειλούνται τα δικαιώματά τους. Άνθρωποι με αναπηρίες δεν είναι παθητικά θύματα, πολέμησαν θαραλέα. Επενεύω την εξαρτία που έχει στην Ιρλανδία κατά περικοπών όσον αφορά εκείνων που παρέχουν περίθαλψη στο σπίτι. Δείχνουν πώ μπορεί να καταπολεθμεί η λιτότητα μέσω μάχη Διασύνδεση με τα συνδικάτα και άλλα κινήματα. Όλα αυτά δεν είναι αναπόφευκτα. Είναι πολιτική επιλογή. Το πολιτικό κατεστημένο σε όλη την Ευρώπη επέλεξε. Τα κατεστημένα επέλεξαν να βάλουν τι τράπεζε, του πλούσιου, του προνομιούχους πάνω από τα άτομα με αναπηρίε. Υπάρχει εναλλακτική που σημαίνει να ξεφύγουμε από τη δικτατορία των αγορών. Που, δηλαδή ότι τεράστιο πλούτο που είναι στα χέρια των μεγάλων εταιριών στην Ευρώπη δεν μπορεί να αγγιχτεί. Αυτό μας λένε. Και το χρέος από εκείνους που έχουν τα μεγάλα ομόλογα πρέπει να πληρωθούν ανεξάρτητο κοινωνικό κόστος. Αυτό πρέπει να το σπάσουμε σαν θέση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα για 1,5 λεπτό δίνουμε το λόγο στην κυρία Γκάλ Πέλτ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Οι κανονισμοί και οι διεθνείς ε, δεσμεύσεις ε, προχωρούν προς τη σωστή κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι μια πολιτική βιτρίνας, διότι η υλοποίηση καθυστερεί και υπάρχουν πολλά κενά. Χρειαζόμαστε μία μεταρρύθμιση της κοινωνικής πολιτικής στον τομέα της πολιτικής της υγείας. Και Μπορώ να μιλήσω για την Ουγγαρία, όπου 14% των ατόμων με αναπηρία δούλευαν πριν από 10 χρόνια, τώρα είναι 13%. Δεν είναι όμως ανταγωνιστικοί οι εργαζόμενοι αυτοί και γι' αυτό θα πρέπει η κυβέρνηση να καταβάλει τις αντίστοιχες παροχές. Θα πρέπει να δίδονται κίνητρα για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία και θα πρέπει να δημιουργηθούν οι δυνατότητες για άτομα με αναπηρία να έχουν ε, πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Και θα πρέπει να υποστηρίζουμε ακόμη και σε διαγωνισμούς ε, τις συμβάσεις που περιλαμβάνουν ε, προϊόντα για άτομα με αναπηρίες. Είναι ιδιαίτερα επίκαιρη η κατάσταση και χρειάζονται συγκεκριμένες λύσεις για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό η κυρία Κοστέλο. Κύριε Επίτροπε, περίπου το 60% του, το 16% συγγνώμη, του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με εμπειρία και το ποσοστό το εργαζομενών ε, ανθρώπων με αναπηρία είναι 45%. Το ποσοστό της ανέχειας μεταξύ ανθρώπων με αναπηρία είναι 17% περισσότερο από το μέσο όρο στην Ευρώπη. Ε, θίγονται οι άνθρωποι αυτοί περισσότερο από τις περικοπές. Κυρίως αυτό ισχύει σε χώρες όπου εφαρμόζονται προγράμματα μεταρρύθμισης όπως η Ιρλανδία, ε, η Τρόικα. Έχει, θέλουμε να ξέρουμε πώ η Κομισιόν μπορεί να διασφαλίσει ότι οι ανάγκε των ανθρώπων με εμπειρία αντικατοπτρίζονται στι κατευθυντήριε γραμμέ για την πρόληψη τη αγωγή διακρίσεων. Πώ θα διασφαλίσει η Κομισιόν ότι τα κράτη-μέρη θα υιοθετήσουν ενεργητικέ πολιτικέ απασχόληση για να βοηθήσουν του ανθρώπου με αναπηρία να παραμείνουν για να μπουν στην αγορά εργασία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πακέτο κοινωνικών επενδύσεων για να μειώσουμε ε, τις ε, διακρίσεις κατά των ανθρώπων με αναπηρία. Έχουμε υποχρέωση να αναλάβουμε άμεση δράση για να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους στην κοινωνία μας και να διασφαλίσουμε ότι, να διασφαλίσουμε ότι γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Ευχαριστώ. Τώρα για ένα μισή λεπτό, κυρία Τζόρνταν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, κύριε Επίτροπε. Ε, τα δικαιώματα σε ίσες ευκαιρίες ε, ε, είναι σημαντικά για την Ευρώπη και αυτό το τονίσαμε και την ημέρα των γυναικών την 8η Μαρτίου. Σε εποχές κρίσης κερδίζει αυτός ο οποίος μπορεί να είναι περισσότερο επιθετικός και μπορεί να ε, αντέχει περισσότερο στις συνθήκες ε, κακουχίας. Και αυτό ισχύει στην αγορά εργασίας, όπου η κατάσταση δεν είναι καλή και προφανώς τα άτομα με αναπηρίες αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι μία από τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η αλληλεγγύη. Η κοινωνία πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματική. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη πειθαρχία. Δεν θα πρέπει να καταναλώνουμε περισσότερα από όσα παράγουμε και θα πρέπει το βάρος να είναι ίσα κατανεμημένο θα πρέπει αυτοί οι οποίοι χρήζουν μεγαλύτερη προστασία να μην είναι αυτοί οι οποίοι επιβαρύνονται περισσότερο από την κρίση. Να δώσουμε μια εγγύηση στου ανθρώπου αυτούς ότι μπορούν να ζήσουν μια ζωή με αξιοπρέπεια. Να, να θέσουμε στόχους ε, για χαμηλότερη ανεργία, για δίκαιη εργασία με ίσε συνθήκε αμοιβή, προώθηση της ε, αλληλεγγύης ε, και κράτος κοινωνικού δικαίου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χόουιτ. Ευχαριστώ. Ε, το ε, Σαββατό ε, διαδήλωσαν κάποιοι άνθρωποι και μας έδειξαν πως οι περικοπές ενός δισεκατομμυρίου του στιγμούν ε, σύμφωνα ε, με το συναπισμό των αναπήρων ατόμων. Ένας στους τέσσερις χάνουν το επίδομά τους ε, και αυτό σημαίνει ότι 6% των γιατρών λένε ότι πολλοί από τους ασθενείς τους ε, προσπάθησαν να αυτοκτενήσουν και ε, τώρα στη δική μου επικράτεια έχουμε 30.000 ανθρώπους να φύγονται από τα οι Άνθρωποι με αποτελούν το 8% του πληθυσμού, αλλά φέρνουν το 29%, υφίσταται το 29% των περικοπών. Στη Βρετανία οι άνθρωποι με ε, δεν υπάρχουν υπηρεσίες για τους ανθρώπους ε, αυτούς για να βγουν από το κρεβάτι, αλλά τους φορολογούν περισσότερο, απλώς επειδή μένουν εκεί και ε, αποσύρεται το επίδομά τους από την κυβέρνηση και οι άνθρωποι με αναπηρίες χάνουν τη βούληση για ζωή. Σας ευχαριστώ και τώρα για μισή λεπτό η κυρία Σταρας Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι επιπτώσεις της κρίσης είναι προφανείς στην κοινωνία στο σύνολό τη, αλλά κυρίως ε, στους πιο ευάλωτες ομάδες όπως στους ανθρώπους με αναπηρία. Έτσι, οι άνθρωποι με αναπηρία μπορεί να ε, να ε, είναι αντικείμενο δευτερογενούς ε, εισαγωγής διακρίσεων. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Ανεπηρία αποτέλεσε ιστορικό μήνυμα. Αυτό δεν αποτελεί το τέλος, αλλά την αρχή μιας διαδικασίας και σύμφωνα με την σύμβαση δεν μπορούμε να επιτρέψουμε μια ομάδα που ήδη ε, δέχεται διακρίσεις ε, να υποστεί διακρίσεις δεύτερη φορά. Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την υπαναχώρηση. Πρέπει όλα τα μέτρα λιτότητας που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη να διατηρούν το επίπεδο προστασίας των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων και τα μέτρα λιτότητα να είναι προσωρινά, αναλογικά και να μην ζημιώνουν σε καμία περίπτωση τα δικαιώματα αυτά τα Ηνωμένα Έθνη έλεγαν ότι σε περίοδους κρίσης οι προσπάθειες ε, πρέπει να διπλασιάζονται για να εγγυόμαστε το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων χωρίς εισαγωγή διακρίσεων και ιδίως των ανθρώπων που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Το άρθρο 27 της Σύμβασης ε, αναφέρεται σαφέστατα στο δικαίωμα της εργασίας, αλλά πριν μιλήσουμε για εργασία πρέπει να μιλήσουμε για συμπεριληπτική εκπαίδευση, όπου όλοι είμαστε ίσοι και να μπορούμε να έχουμε τις ίδιες ευκαιρίε. Έτσι λοιπόν ζητώ από την Κομισιόν και την Επίτροπο να συνεχίσει στην οδό αυτή για να μπορέσει να ζητήσει από όλα τα κράτη-μέλη τα λιτότητα, η λιτότητα και τα μέτρα λιτότητα να μην ζημιώνουν του ανθρώπου με αναπηρία. Ευχαριστώ και τώρα κυρίε και κύριοι. Έχουμε τη διαδικασία Catch τη αλλά θα ήθελα να σας πω ότι 12 άτομα έχουν ζητήσει το λόγο και η διαδικασία προβλέπει μόνο 5 λεπτά και ο συνολικός ε, χρόνος για τη συζήτησή μας ήταν μέχρι τις 11 και έχουμε καθυστερήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι θα δεκτώ να πάρω το λόγο όσοι δεν είχαν να μιλήσει στο παρελθόν. Η κυρία Τσελέσκα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δύσκολο αυτό το θέμα είναι σημαντικό και θα ήθελα να πω ότι πράγματι πρέπει να δείξουμε στους πολίτες ότι δεν δεχόμαστε τον αποκλεισμό των ομάδων αυτών των ανθρώπων με αναπηρίες. Δυστυχώς σε μια περίοδο λιτότητας αυτό είναι κάτι που εμφανίζεται. Θα πρέπει να σκεφτούμε την κινητικότητα και των ατόμων με αναπηρία ούτω ώστε αυτά τα άτομα να μπορούν να συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας. Και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες. Όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει στις εργασίες τους ε, να λαμβάνουν υπόψη ε, το θέμα της ίσης μεταχείρισης και να έχουν αυτό το στόχο ε, στις πολιτικές τους. Κάνω μια έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κράτη-μέλη θα πρέπει να βρουν τις κατάλληλες λύσεις ε, ούτω ώστε να μπορέσουν τα άτομα με αναπηρία να ζουν μια αξιοπρεπή ζωή. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία θα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Εμεί στην Ιρλανδία έχουμε μισή δεκαετία λιτότητα όταν σχεδόν ε, κατέστραφε όλο ο χρηματοπιστωτικό ε, τομέα στον κόσμο και αυτοί που στην εξουσία αποφάσισαν να τον σώσουν με ει βάρο των πολιτών και των προλογωμένων. Η λιτότητα θεωρείται ότι είναι ε, τελικά ένα μέσο για να γλιτώσουν χρήματα. Αυτό επιβάλλουν. Θα μπορούσα να δώσω πολλά παραδείγματα στον Επίτροπο Ρεν που τελικά ε, προσπαθεί να κατεβάσει τις προβλέψεις, θα ήθελα να του πω να έρθει να δει στην εκλογική περιφέρεια αυτά τα μέτρα του τι κάνουν στους ανθρώπους με πραγματική ανάγκη. Και το πείδωμα ανεργία στην Ιρλανδία επέτρεπε στον κόσμο να ζήσει με ανεξαρτησία και να είναι ενεργό στην κοινότητά του. Και αυτό πρόκειται να διακοπεί σε τέσσερι μήνε. Και δημιουργείται ερωτηματικό, ποιο μελλοντικό σχήμα θα αντικαταστήσει αυτό. Η χρηματοδότηση για υπηρεσίε που παρέχονται οι ηλικιωμένου στο σπίτι είναι κάτι που χρηματοδοτείται λιγότερο. 14% από, 40% από του ηλικιωμένου δεν έχουν καμία υποστήριξη και διδασκαλία με παιδιά που έχουν προβλήματα μάθηση τα επιδόματα σχετικά έχουν μειωθεί. Και τελικά έχει μειωθεί η υποστήριξη. Θα εκτιμούσα να ακούσω κάποια απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σα ευχαριστώ που μου δώσατε το χρόνο. Και τώρα, για ένα λεπτό, ο κύριος Σόγκορ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι αρνητικές ε, συνέπειες οξύνθηκαν λόγω των μέτρων ε, λιτότητας. Αυτά τα μέτρα λιτότητας ε, πλήττουν ιδίως τα στρώματα της κοινωνίας που χρειάζονται μεγαλύτερη προστασία. Καλό θα ήταν να μπορέσει να δώσει συστάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να προτείνει και βέλτιστες πρακτικές προς τα κράτη-μέλη προς την κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσουν για να ενισχύσουμε την απασχόληση για τα περισσότερο αδύναμα άτομα. Ξέρουμε ότι στα νέα κράτη-μέλη είναι χειρότερες οι συνθήκες από ότι στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για τις χώρες αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Νικολάσικ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Οι λιγότερο εκπαιδευμένοι άνθρωποι, οι ευάλωτοι άνθρωποι, εκείνοι που διατρέχουν τον κίνδυνο αποκλεισμού, οι άνθρωποι με αναπηρίες και κυρίως με συνδυασμένη αναπηρία και φυσική και ψυχική είναι οι πιο ευάλωτοι άνθρωποι που κατά τη διάρκεια μιας περίοδου κρίσεως μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να είναι οι πρώτοι στόχοι, να είναι τα πρώτα θύματα, αυτοί που θα χάσουν τη δουλειά τους, οι πρώτοι άνθρωποι που θα μπουν στη φτώχεια. Σε άλλες περιόδους, χωρίς κρίση, και πάλι αυτοί οι άνθρωποι είναι στο περιθώριο όσον αφορά τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Και χαίρομαι που τώρα στις 11 και 20 το βράδυ ακόμα συζητούμε αυτό το σημαντικό θέμα παρά το προκεχωρημένο της ώρας. Εκτιμώ τα όσα είπε η κυρία Επίτροπος. Είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει τη σύμβαση για τις αναπηρίες και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να βρει τρόπους ώστε να προσέξει αυτά τα άτομα. Ο παπα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώ η κρίση, και αυτό το γνωρίζουμε πολύ καλά, ιδίω στι χώρε με τα μεγαλύτερα προβλήματα, όπω η Ελλάδα, δεν κάνει διακρίσει. Και αναφέρθηκε προηγουμένω και η κυρία Επίτροπο στα προβλήματα των χωρών αυτών. Δεν διακρίνει τα άτομα που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη την κοινωνική προστασία. Δεν διακρίνει εκείνου που τι δύσκολε ώρε η στήριξή του είναι περισσότερο επιτακτική. Θα αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα από την Ελλάδα το ποσοστό ανεργία σήμερα ανέρχεται κοντά στο αβάστακτο 27%. προσέξτε όμως η ανεργία των ατόμων με ειδικέ ανάγκες ξεπερνάει το 55% φτάνει δηλαδή στα επίπεδα της ανεργία των νέων. αν επομένω για κάποιον μέσα στην κρίση είναι δύσκολο να βρει εργασία για έναν συνάνθρωπό μας που αντιμετωπίζει για παράδειγμα κινητικά προβλήματα αυτό είναι σχεδόν αδύνατον σωστά αναφερόμαστε και το κάναμε και σήμερα σε ζητήματα περίθαλψης σε ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας είναι απόλυτα αναγκαίο θα πρέπει όμως να δούμε και θέματα πρακτικά όπως η εργασία που πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί έχουν εξαιρετικές δεξιότητες και μπορεί να αποβεί προς όφελος και των ίδιων αλλά και των κοινωνιών τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τζούμπερ είναι τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ. Στην Πορτοβαλία τα άτομα με αναπηρία αποτελούν περίπου ένα εκατομμύριο οι εθνικέ οργανώσει ατόμων με εμπειρία έκαναν ανάλυση των επιπτώσεων ε, των μέτρων που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και κατέληξαν στο ότι υπάρχει περισσότερη ανέχεια και κοινωνικό αποκλεισμό που πλήττουν περισσότερα τα άτομα με αναπηρίε και έχουμε πολλαπλέ περιπτώσει έλλειψη πρόσβαση σε υπηρεσίε υγεία και υπάρχει μεγαλύτερη έλλειψη πρόσβασης σε φάρμακα και υπάρχει πολλές φορές αδυναμία να μπουν οι άνθρωποι αυτοί στην αγορά εργασίας και κάθε φορά ε, υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις ε, πείνας και υποσυτισμού. Τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υποστήριξα να πω τις μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες αυτού του Κοινοβουλίου έχουν ε, τελικά οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση τα άτομα είναι πύροι. Η Ευρώπη είναι ε, μια Ευρώπη καλών προθέσεων, όμω τελικά οδηγεί του ανθρώπου αυτού σε μια δεινή κατάσταση, σε απάνθρωπη κατάσταση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πρέπει να κλείσω αυτή τη διαδικασία κατσδιάη. Ξέρω ότι θα θέλετε να διαμαρτυρηθείτε, αλλά λυπάμαι πολύ. Εγώ σεβόμαι όλου τους κανόνες εδώ. Θέλω να δώσω το λόγο στην κυρία Ρέντινγκ για να ολοκληρώσει, να κάνετε τελικά τη σχόλια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τους ανθρώπους με αναπηρία και θα την γνωρίζετε πολύ καλά γιατί ε, ισχύει από το 2010 βοηθά τα κράτη-μέλη να προωθήσουν την κοινωνική ένταξη και ακόμη και αν τα κράτη-μέλη είναι αυτά που είναι βασικά αρμόδια ε, για τους τομείς της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθά τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε αυτό το τομέα αν δούμε για παράδειγμα το ποσοστό της απασχόλησης με δράσεις όπως η απασχόληση ατόμων με αυτισμό και άλλες διαταραχές. Έχουμε ε, ειδικό πρόγραμμα για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να βοηθήσουν ε, τους ανθρώπους αυτούς ε, να ενταχτούν σε προγράμματα εργασίας ε, και η Κομισιόν προσπαθεί να βρει λύσεις και βέλτιστες πρακτικές για τα κράτη-μέλη για πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Όμως βέβαια η Κομισιόν πρέπει να συνεισφέρει και η ίδια από μόνη της. Και ο συνάδελφος Άντορ παρουσίασε το πακέτο κοινωνικών επενδύσεων που χρησιμοποιεί η Κομισιόν προκειμένου να καθοδηγήσει τα κράτη-μέλη να επενδύσουν ε, τους απαραίτητους πόρους ε, πιο αποτελεσματικά για την προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της κοινωνικής συνοχής. Η στρατηγική, όπως ε, ρώτησε ο κ. Κόζα, θα αναθεωρηθεί φέτος και θα δημοσιευτεί και μία έκθεση για την εφαρμογή της στρατηγικής θα δοθεί στο κοινοβούλιο το εγγραφό αυτό με τα θετικά στοιχεία, αλλά θα αναφέρουμε και τι δεν καταφέραμε να κάνουμε. Και όταν λέω εμείς, εννοώ την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Όμως, αυτό που κάνουμε είναι να επαναδιοχετεύουμε τα ταμεία, τα κονδύλια των διευθυντικών ταμείων, ε, όχι μόνο τα σημερινά, αλλά και τα αυριανά. Γιατί στο ρυθμιστικό πακέτο των διαφορετικών ταμείων για το 2014-2020, προσδιορίσαμε ε, αρκετά του τομεί ε, που αφορούν την αντιμετώπιση των αναγκών ατόμων με αναπηρία. χάρι χάρη μετάβαση από ε, την θεσμική, συγγνώμη, την ιδρυματική σε ε, περίθαλψη που θα βασίζεται στην κοινότητα. Έτσι λοιπόν θα υπάρχει και μια πρόταση σχετικά επιτάπητος. Τα διαφορετικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βοηθούν τα κράτη-μέλη στους τομείς και τα μοντέλα πρόσβαση σε προσωπική βοήθεια υπάρχουν μέσα στρατηγική και αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τέτοιες δράσεις. Και είπα και το εννοώ ότι πρέπει να υιοθετήσουμε μια διαφορετική άποψη ως προς την προώθηση των υπηρεσιών σε αυτούς τους τομείς, γιατί ε, έχουμε γυράσκοντα πληθυσμό και θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από υπηρεσίες. Και επίσης ε, ένα φάσμα διαφορετικών επαγγελμάτων μπορεί να δημιουργηθεί. Θα ζητήσω από τα κράτη-μέλη οι θέσεις αυτές εργασίας ε, να συμβάλλουν στην ανάπτυξη. Θα είναι σημαντικές θέσεις εργασίας, όχι ίσονος Ευχαριστώ κύριε Συγήτρια που καταδείξατε αυτό το πολύ δύσκολο ζήτημα και ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους σε αυτό τον Νίκο που πήραν το λόγο. Η Κομισιόν θα συνεχίσει να εργάζεται για τα θέματα αυτά με τη δική σας αρρωγή. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Ευχαριστώ όλους τους αγορητές. Ευχαριστώ τους διερμηνείς. Πέρα στις συζητήσεις. Η επόμενη συνεδρία θα λάβει χώρα Άταρτη, 13 του μήνος, από τις 9 μέχρι τις 2 το μεσημέρι και το απόγευμα από τις 3 μέχρι τις 11 το βράδυ. Διαδικαστικό, ορίστε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Διαδικαστικό. Θα προσέξατε το προηγούμενο ότι ζητούσατε δικαστικό. Και το έχω ξαναπεί, όταν ο Πρόεδρο βλέπει ένα μέλο που θέλει να μιλήσει για διαδικαστικό, πρέπει ο Πρόεδρο να το δεχτεί το διαδικαστικό. Ήσασταν εκτό των ε, ευθυνών σα που δεν με είδατε πριν. Το διαδικαστικό